Ε, θέλω να αναφερθώ εδώ εις ε, την, ε, το ναυάγιο κοντά στη Σικελία και δίνω το λόγο τον Επίτροπο Μπαρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε με λύπη την, το ναυάγιο στη, την Κυριακή το βράδυ ε, μίας, ε, ενός σκάφους με 257 άτομα που επέβαιναν εκ των οποίων οι περισσότεροι χάθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εκφράσει την λύπη της ε, για αυτή την ανθρώπινη καταστροφή και το θυμό της διότι οι λόγοι του δράματος αυτή είναι πολλαπλοί και ουσιαστικά οφείλονται εις τις εγκληματικές οργανώσεις που κατευθύνουν απευθύνουν από την Λιβύη αυτή την θανατηφόρα δραστηριότητα και πλουταίνουν μέσω αυτής της οδού. Είναι κρίμα ότι όλα αυτά συνεχίζουν να αναπτύσσονται και ε, καλή επιτροπή όλους να προσπαθήσουν να σταματήσει αυτό το εμπόριο. Η Λιβύη εδώ πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να δεσμευτεί πιο αποφασιστικά και πιο αποτελεσματικά να κατα πολεμήσει τις ε, διακινήσεις αυτές ε, επί του εδάφη τους διότι παράνομες ε, αναχωρήσεις από τις ακτές της θα πρέπει να επιληθούν με την φρούρηση των υδάτων που είναι τα χωρικά της είδητα της βοηθείας προς τα άτομα που χρειάζονται σύμφωνα με την συνθήκη, ε, την Παναφρικανική συνθήκη του 1969 για τους πρόσφυγες την οποία έχει προσυπογράψει. Ε, χρειάστηκε επανειλημμένος να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Λιβύη να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναλάβει αποτελεσματικά μέτρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Πρέπει να σας πω ότι προτείναμε μια οικονομική βοήθεια συνεχώς αυξανόμενη προς τη Λιβύη. Αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει οι αρχές της Λιβύης να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βοήθεια για να βελτιώσουν την καταπολέμηση της διακινήσεως αυτής των προσφύγων και για ενισχύσουν τους ελέγχους των νοτίων ε, συνόρων τους. Θα πρέπει επίσης να δέχονται τους πρόσφυγες σεβόμενοι τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να συμβάλλει εις ε, την σύλληψη και, ή ε, στη βοήθεια των πλοίων αυτών στην Μεσόγειο και στις επόμενες μήνες θα αρχίσουν οι επιχειρήσεις ναυτίλος και ερμής που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της Frontex και θα κοστίσει περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ. Όντως ε, ισχύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν ή στην εφαρμογή εφαρμογή αυτών των δύο δράσεων και θα χρειαστεί επίσης τα κράτη-μέλη να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους συγκεκριμένα προς την Ιταλία και τη Μάλτα οι οποίες εκτίθενται πάρα πολύ ε, τις μετακινήσεις αυτές από τη Λιβύη και η Λιβύη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για να μπορέσει να αναλάβει και πάλι τους μετανάστες αυτούς οι οποίοι διέρχονται από τα εδάφη της. Έχουμε σημειώσει ότι οι αρχές της Ιταλίας πίστευαν ότι θα ήταν δυνατόν από τις 15 Μαΐου να υπάρξουν ε, κοινέ ε, περιφρουρήσεις των ε, υδάτων της Λιβύης μαζί με τους Λιβύους για να μπορέσουν να συλλαμβάνουν και να σταματούν αυτά τα παράνομα φορτία και ε, στηρίζουμε τις, ε, τη βοήθεια της ε, Ιταλίας προς την αδευτική δύναμη της Λιβύης με αυτό το στόχο. Θεωρούμε όμως ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει συγχρόνως η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος διότι οι ε, μετανάστες οι οποίοι αναθέτουν τη ζωή τους εις ε, τους λαθρεμπόρους ε, διαφεύγουν από κινδύνους ή φυγαδεύονται και τα γεγονότα αυτών των τελευταίων ημερών σε όλα τα κράτη-μέλη ε, μας οδηγούν στο να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος κατά τρόπον ώστε μαζί με τα κράτη-μέλη και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος των προτεραιοτήτων του σε αυτή την γενική προσέγγιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται μία συνολική προσέγγιση για να εκπονηθεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για να λάβει υπόψη ε, τις ε, ροές των μεταναστάσεων, να λάβει υπόψη το, τις χώρες προελεύσεως και από την άλλη πλευρά η στρατηγική αυτή θα πρέπει να επιτρέψει να εμβαθύνουμε την συζήτηση που έχουμε και το διάλογο με τις χώρες της Αφρικής στα πλαίσια της διαδικασίας του Ραμπάτ στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Αφρικανικής Ενώσεως. Από κοινού θα πρέπει να εντοπίσουμε κοινέ απαντήσεις για να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτές και επίσης θα πρέπει να επωφεληθούμε των ευκαιριών που δίνει μία τακτική μετανάστευση που μπορεί να είναι μία ευκαιρία και για την Ευρώπη και για τις χώρες αυτές προελεύσεως. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να κινητοποιήσει επιπρόσθετους πόρους και να εντείνει την συνεργασία με τις χώρες προελεύσεως και διελεύσεως να ενισχύσει τη δυνατότητά τους να διαλύσουν ε, τις ε, της ε, οργανώσεις αυτής των λαθρεμπόρων και να συμπεριφέρεται προς τα άτομα αυτά σεβόμενοι τον νόμο. Θα πρέπει συγχρόνως να οργανώσουμε την άφηξη των ατόμων αυτών που ζητούν νόμιμα άσυλο να μπορέσουμε καλύτερα να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, πριν από 15 μέρες πήγα στη Λαμπεντούζα και στη Μάλτα. Πρέπει να σας πω ότι διαπίστωσα η διεισόμαση και άκουσα τα δράματα των ατόμων αυτών που έχουν ε, κληθεί από λαθρεμπόλους ε, να ε, περάσουν προς την Ευρώπη με κίνδυνο της ζωής τους. Κατόπιν λοιπόν αυτού του τελευταίου γεγονότος θα πρέπει να θεωρήσουμε τα προβλήματα αυτά ως πάρα πολύ σοβαρά και να ζητήσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιηθεί η σοβαρότης και ε, η επιτάχυνση αυτού του φαινομένου που θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή υπό φρικτές συνθήκες. Γι' αυτό και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ζητά από την Επιτροπή αυτή την δήλωση την οποία προσφέρω δηλώνοντας πολύ συνειδητά ότι στους επόμενους μήνες θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποφύγουμε τέτοιες και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε ε, Επίτροπο, κύριος Διάς Δεμέρα για δύο λεφτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σήμερα συνειδητοποιήσαμε συλλογικά για τον πόνο και την αλληλεγγύη για τον θάνατο στη Μεσόγειο τόσων μεταναστών που ήταν απεγνωσμένοι και με τόσες ελπίδες αλλά και απογοητεύτηκαν και βρέθηκαν σε απόγνωση. Είναι αθώα θύματα και που δεν επέλεξαν αυτούς τους όρους που τους επιβλήθηκαν και αυτές τις καταστάσεις. Γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα. <clears throat> Στην Μεσόγειο και στην ακτή του Ατλαντικού για πολλούς που δεν έχουν τίποτα πια στον κόσμο υπάρχει η χρυσή οδός προς το χρυσό μέλλον στο Ελντοράδο και έτσι εδώ όταν φτάνουν ε, στην, ε, ε, στον προορισμό τους αυτά όλα απογοητεύονται. Πρέπει να είναι πολύ πιο ευαίσθητη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφεύγουμε τέτοιες τραγωδίες. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σκληρά και ομά όπως είδαμε και στις ακτές της Λιβύης. Πρέπει αυτό να μας κάνει να σκεφτόμαστε την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια και συνταγές για να υπάρξουν ε, <clears throat> απόλυτα αποτελεσματικές ε, πολιτικές ε, λύσεις για το δράμα. Όμως πρέπει να έχουμε βιώσιμες πολιτικές. Πρέπει να διατηρήσουμε πολιτικές αλληλέγγυες σε συνεργασία με τις χώρες διαμετακόμισης και προέλευσης και να δούμε για τη μετανάστευση τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Πρέπει να μπορέσουμε καλύτερα την νόμιμη μετανάστευση να τη διαχειριστούμε με τα προτερήματα που συνεπάγεται ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις χώρες προέλευσης και διαμετακόμψης στους ελέγχους των συνόρων και πρέπει να ε, με συνετό και εφάνταστο τρόπο να καταδιώκουμε εκείνους που είναι λαθρέμποροι ανθρώπων και να εφαρμόζονται οι ποινικέ διατάξεις. Πρέπει καλύτερα να εξοπλίσουμε το Ταμείο Φύλαξης Εξωτερικών Συνόρων. Ένα 1.800 ε, εκατομμύρια για μεγαλύτερη χρονική περίοδο είναι ένα επαρκές ποσό. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τη Frontex. Ο κατάλογος ε, των μέσων σε σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν να μην είναι ένα ευχολόγιο, αλλά να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να συντονίζουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα κομβικά σημεία. Στα κομβικά σημεία μεγαλύτερης πίεσης, ιδιαίτερα παράνομης μετανάστευσης πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με τα όσα ε, ε, αναφέρονται σε αυτά τα ποσά συμβάλλουν με μεγαλύτερη δέσμευση για την αύξηση των προσπαθειών. Πρέπει να πάψουμε να κάνουμε διακηρύξεις και πρέπει να περάσουμε στις πράξεις ώστε να εστιαστούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να επομιστούμε τις σκληρές ε, τις ομές, με ομό τρόπο τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εδώ μιλάμε για την εξαφάνιση χιλιάδων ειδών. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται. Μερικές χώρες σαν την Ιταλία υπογράφουν διμερείς συμφωνίες όπως τη σύμβαση που υπέγραψε πρόσφατα με την Λιβύη η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από την απικιακή ήδη εποχή και κάνει παραχωρήσεις για να ελεγχθεί κάπως η μεταναστευτική ροή από εκεί. Έρχονται από την Ευρώπη, ας πούμε, για τη Λιβύη από την Ιταλία, χιλιάδες νέοι των οποίων φυσικά τα όνειρα καταστρέφονται και τα γαλλικά συμφέροντα στον Ήγυρα το ίδιο φαινόμενο δημιουργούν ε, για την εκμετάλλευση του ουρανίου. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος μεταξύ του ΑΡΕΓ γιατί έτσι εποφελούνται όλοι αυτοί οι δουλέμποροι και το βλέπουμε και από τον τύπο ακόμη. Άρα ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίζουν με τη φωτιά και αν δεν αλλάξει αυτή η στάση σύντομα, αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει να αντιδράσει με θετικά και συνεπή προγράμματα που να συμφωνούν με τις αρχές μας, τότε δεν θα αρκέσει πια να αποσιωπούμε τα γεγονότα όπως γίνεται τελευταία, αλλά θα γίνει φανερό ότι η Μεσόγειος τελικά είναι ένα, θα γίνει ένας τεράστιος ε, τάφος. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα λάβει το λόγο για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες ε, για την Ευρώπη. Ε, ένα λεπτό, κύριος Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, και εγώ εν ονόματι της η ομάδος μου υποκλίνομαι εις το γεγονός αυτό αλλά δεν φτάνει η συμπόνια πρέπει να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο την πραγματικότητα δηλαδή ότι τα πραγματικά νότια σύνορα της Ευρώπης δεν είναι στην Ευρώπη αλλά στην ε, Αφρικανική Ήπειρο μόλις ε, ε, φύγουν ε, τα πλοία από τις ακτές της Αφρικής δεν υπάρχει για τους επιβαίνοντας καμία επιλογή είτε θα αποπευθούν εάν φτάσουν στην Ευρώπη είτε θα υποκύψουν καθοδόν. Μόνο όταν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με τις χώρες προελεύσεως και διελεύσεως πραγματικά πραγματικές συνεταιρικές σχέσεις θα μπορέσει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος των συνόρων και ιδέως μία ουσιαστική προσφορά για νόμιμη μετανάστευση και ε, για ουσιαστική βοήθεια προς την ανάπτυξη. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα θαλάσσια ατυχήματα παρόλη ε, την ε, συμπόνια την οποία εκφράζουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέ για τους πράσινους και την συμμαχία τους δυόμιση λεπτά η κυρία Φλότρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ποιοι ήταν, πόσοι ήταν, υπήρχαν παιδιά, γυναίκες, πρόσφυγες. Οι ακτοφύλακες εμπόδισαν ε, να περάσει το, ε, το πλοίο, οι αλλοί του είδαν, δεν γνωρίζουμε, αλλά εκατοντάδες χάθηκαν και έρχονται να αυξήσουν τις χιλιάδες που έχουν χαθεί στην Μεσόγειο ή ε, να καταλήξουν ε, σε ε, εξορία υπό απάνθρωπες συνθήκες γιατί φεύγουν από κατεστραμμένες περιοχές, δεν έχουν άλλες διεξόδους και αυτοί είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν τους μετανάστες να χρησιμοποιήσουν συνέχεια πιο επικίνδυνες δρόμους διότι στις επόμενες μέρες ανακοινώνονται αυτές οι ε, κοινέ περιπολίες της Ιταλίας και της Λιβύης και γι' αυτό βιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν προς την Ευρώπη και να χρησιμοποιήσουν τη θανατηφόρα αυτή μέθοδο τα συρματοπλέγματα και οι περιπολίες δεν τους εμποδίζουν να διαφύγουν. Άρα το ερώτημα είναι η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει τις επιπτώσεις μιας τέτοιας επιλογής. Δεν το γνωρίζουμε και γι' αυτό παρακαλώ την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσουν τα άτομα τα οποία χάθηκαν και να ερευνήσουν τις συνθήκες αυτού του ναυαγίου, να προσαρμόσουν το δικαίωμα της θαλάσσης που ζητά ε, να ε, βοηθηθούν ε, οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης υπάρχουν συνεργασίες με χώρες που δεν σέβονται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να, τα άτομα αυτά και οι πρόσφυγες να μπορέσουν να διαφύγουν προς οποιαδήποτε χώρα. Δεν πρόκειται για παράνομο νόμους ε, μετανάστες. Πρόκειται ε, για αυθαίρετες κρίσεις και θα πρέπει να αναπτυχθεί η ανθρώπινη πολιτική στις τρίτες χώρες ε, της Αφρικανικής Υπήρου μέσω όλων των δυνατών δυνατοτήτων ακόμη και αν χρειαστεί να συνεργαστεί κανείς με τους δικτάτορες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την Ανατολική Αριστερά. Για δυόμιση λεπτά ο κύριος Κατάνια παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το οποίο συνέβη προχθές είναι το τελευταίο δράμα, η τελευταία, το τελευταίο γεγονός που μας ντροπιάζει και που έχει μια πραγματικά ανευπροηγουμένου ε, διάσταση Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραβίαση στο δικαίωμα στη ζωή στην ίδια την Ευρώπη. Αυτό το δράμα δείχνει ότι το φρούριό μας ε, δεν ε, βαίνει καλώς ε, και πρέπει να... Σε αυτό οφείλεται αυτή η εσχήνη τα θύματα αυτά, γυναίκες και άνδρες που ήθελαν να ζουν καλύτερα και προσπάθησαν να ξεφύγουν από την πείνα και από τον πόλεμο, οφείλονται σε αυτό το φρούριο, το έσχος δεν είναι απλά μια ανομαλία, μια κατάσταση που δημιουργεί παράνομη μετανάστευση. Είναι μια προβλέψιμη συνέπεια της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά συμβαίνουν στη Μεσόγειο λόγω της καταστολής και λόγω της καταδίωξης ε, στη θάλασσα. Τα όσα γίνονται στις ακτές μας, απαγορευτική πολιτική των κρατών μελών καταστολή και εις βάρος αυτών των μεταναστών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσουν στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν διάβλοι ώστε να μπορέσουν με διαφορετικό νόμιμο τρόπο να καταλήξουν στην Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι και παραβίαση των ιερών δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. Και όλα αυτά διαδραματίζονται στην Μεσόγειο. Και οι διοκτήτες αυτών των πλοιάριων και πλοίων εκμεταλλεύονται με κάθε τρόπο και ανελέητα τις ε, διάβλους ε, προς την Ευρώπη. Αυτοί είναι στους οποίους οφείλονται αυτά τα θύματα. Για παράδειγμα πρόσφατα στις ακτές της Λιβύης. Οι ε, μετανάστες που πέθαναν, αποβίωσαν είναι μυριάδες μπορούμε να πούμε κατά τα τελευταία χρόνια γυναίκες και άνδρες που απεβίωσαν στη θάλασσα με ένα λεπτό σε αυτή την ε, σύνοδό μας, σε αυτή την ολομέλεια, θα πρέπει να ποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτά τα άτομα. Ως ελάχιστη απότιση φόρου τιμής προς, αυτά τα, προς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ για την ε, αποδοχή της, ε, του αιτήματό μας. Δεν επαρκεί όμως αυτό. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη χειροπιαστή πολιτική για να πούμε και να, από αυτό το κοινοβούλιο ποτέ ξανά να μην υπάρξουν θύματα στη Μεσόγειο. Σα ευχαριστώ. Στην συνέχεια θα λάβει τον λόγο επίτροπος Μπαρό, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Αυτό που έχει σημασία είναι να δράσουμε. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο πρόεδρος Ντεπρέ. Πρέπει όντως να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, συνολική προσέγγιση και την εταιρική, τις εταιρικές συμφωνίες διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε λύσεις. Όπως είπατε έχουμε σαν Ευρωπαίοι ευθύνε. Πρέπει αφενός όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση να είμαστε ανοιχτοί. Θα πρέπει επίσης να, ε, να λάβουμε τις ευθύνες μας για την ε, ανάληψη και την υποδοχή των ατόμων που διαφεύγουν στον πόλεμο αλλά όπως λέγεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σωστά ε, δυστυχώς υπάρχουν και ορισμένα κράτη τρίτα με τα οποία είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς. Πρέπει όμως να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Όχι. Η Λιβύη θα πρέπει να έχει ένα σύστημα ασύλου. Θα πρέπει η Λιβύη να μπορέσει να μας βοηθήσει να σταματήσουμε ορισμένους λαθρεμπόρους οι οποίοι αναλαμβάνουν φοβερές, ε, φοβερούς κινδύνους και θέτουν σε φοβερό κίνδυνο αυτά τα άτομα και οι αρχές της Μάλτας μου έχουν πει ότι η Λιβύη αφήνει και να αποπλέψουν πλοία σε τραγική κατάσταση και μετά η ε, ναυτιλία της Μάλτας είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει να βοηθήσει ε, και να σώσει τα άτομα αυτά που εκμεταλλεύονται οι λαθρέμποροι. Βεβαίω θα πρέπει όμως σε όλα αυτά να είμαστε στεναροί και στις διαπραγματεύσεις για τα κράτη που δεν αναλαμβάνουν και δεν σέβονται τις, εθνικές, τις διεθνείς τους ευθύνες. Θα πρέπει όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την επιστροφή τέτοιων δραματικών γεγονότων. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Λάξ για τον κοινοτικό κώδικα θεωρήσεων διαβατηρίων. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Λάξ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε